Περνώ στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι το θέμα του, της οργάνωσης Boko Haram και δίνω το λόγο στους ομιλητές κύριο Κριστιανό Πρέντα καταρχάς για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πριν από ένα χρόνο ακόμα μιλούσαμε το θέμα των ε, φρικαλαιοτήτων της Μπόκο Χαράμ στην Ιγυρία. Δυστυχώς έχει περάσει ένας χρόνος και τίποτα δεν άλλαξε. Συνεχίζονται οι ένοπλες επιθέσεις, οι ε, δολοφονικές επιθέσεις, οι απαγωγές από την Μπόκο Χαράμ ε, και, μάλιστα έχουν πολλαπλασιαστεί. Πρέπει να τι καταδικάσουμε λοιπόν απερίφραστα. Ταυτόχρονα πρέπει να ζητήσουμε την άμεση αποελευθέρωση των κοριτσιών που απήχθησαν από το σχολείο του στο Σίμποκ και να, στήσουμε την, ε, και να καταδικάσουμε μαζί με τη διεθνή κοινότητα την ε, οργάνωση αυτή. Ιδιαίτερα καταδικάζουμε δε την ε, προώθηση των, του, της τζιχάτ και των Ισλαμιστικών ακρεωτήτων τόσο στην Ιγυρία όσο και στη Σομαλία από ομάδες τρομοκρατικές οι οποίες αποτελούν απειλή για την ίδια τη ζωή και την ασφάλεια οποιοδήποτε δεν ενστερνίζεται τις δικές τους απόψεις. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια μεγάλη απειλή τη σταθερότητα της χώρα και για την ευρύτερη διότι βεβαίω καταδικάζουμε κάθετα όλε αυτέ τι βιότητε ε, που κάνει η μου και τις πράξεις κατά των πολιτών και έχουμε πάνω από 270 μαθήτριες από το ε, σχολείο του Τσίμποκ. Οπότε όλα αυτά θα πρέπει να κατηγηθούν στη δικαιοσύνη. Δεν θέλουμε η Μποκοχαράμου να ενωθεί με άλλες συμμορίες και με εμπόριο ναρκωτικών. Ε, θα πρέπει να δώσουμε μια απάντηση αποτελεσματική. Η ιδέα διακηρύξεις μας να δούμε το ότι δεν αρκούν. Θα πρέπει να συνδυάσουμε την ασφάλεια με μια πολιτική ανάπτυξη και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτική για την παιδεία, καταπολέμηση της διαφθοράς, συνεργασία σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο για να καταπολεμήσουμε αυτές τις συμμορίες, αλλά όμως ποτέ δεν θα έχουμε μια αυθεντική εξωτερική πολιτική από πλευράς Ευρώπης εάν δεν υπάρξει στρατιωτική δυνατότητα όταν χρειάζεται η άσκηση βία. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος και τώρα ο κύριος ε, Τάνο για 1,5 λεπτό. Πρόκειται για αυτές τις ε, αποτρόπες ε, επιθέσεις γιατί 44 φώνευσαν και έκαψαν τρεις εκκλησίες σε κάποιο χωριό της Μποκαχαράμ θεωρούν ότι η δυτική παιδεία είναι αμάρτημα και θεωρούν ότι οι θρησκευτικέ μειονότητε και ιδίω οι χριστιανοί επίση είναι εγκληματίε. Πρόκειται για όλο το Σαχέλ όπου έχει χτυπήσει αυτή η, η τρομοκρατία στην Μέση Ανατολή και στη Σομαλία και ακόμα και μέχρι το Αφγανιστάν και το Πακιστάν υπάρχει τέτοια τρομοκρατία από τους Ταλίμπα. Τώρα θα πρέπει μαζί με τις ΙΠΑ ε, ε, να αντιμετωπίσουμε αυτή την απειλή και με την Ρωσία και με την Κυριακή με την Ινδία γιατί όλοι Έχουμε συμφέρον το πολεμήσουμε την πολιτική τρομοκρατία και θα πρέπει αυτό το φαινόμενο να αντιμετωπιστεί σφαιρικά και όχι περιπτωσιολογικά. Είδατε τι έγινε στην Νιγηρία. Ε, υπάρχει φτώχεια, οι περισσότεροι ζουν με ένα δολάριο την ημέρα και όλοι αυτοί εκμεταλλεύονται τη φτώχεια ε, και το ότι ο κόσμος δεν έχει δουλειά και φαγητό. Οπότε θα πρέπει να δούμε ότι είναι ενδυμικό φαινόμενο η διαφθορά δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους η, η, η αστυνομία και άλλες αρχές. Σας ευχαριστώ λοιπόν και διακόπτω. Δυστυχώ μέχρι τώρα η απόκριση μα ήταν ανεπαρκή Παρακαλώ, συνάδελφοι, λέει ο πρόεδρο, καθίστε, κάντε ησυχία να συνεχιστεί η συζήτηση. Η κυρία Τζιν Λάμπερτ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι στις αρχές του έτους ε, είδαμε με μεγάλη, μεγάλο αποτροπηγισμό τις απαγωγές ε, των κοριτσιών και είδαμε την αντίδραση της κοινωνίας στην Ιγυρία. Οι άνθρωποι που στηρίζουν την εκπαίδευση των αγοριών και των κοριτσιών για αυτούς οι επιθέσεις ε, της Μποκοχαράμ δεν είναι μόνο επιθέσεις εναντίον των κοριτσιών. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν την αλλαγή στην Ιγυρία, δράση κατά της Μπόκο Χαράμ, την ανάληψη ευθυνών από την κυβέρνηση και την καταδίκη όλων αυτών που είναι υπεύθυνοι για τις ε, βιοπραγίες. Εμείς λοιπόν εκφράζουμε τη συμπάθειά μας ε, για τις οικογένειες, όχι μόνο των απαχτισών ε, κοριτσιών, αλλά όλων εκείνων διαφορετικής θρησκείας που απήχθησαν, που δολοφονήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των ετών με την αυξανόμενη βία της Μπόκο Χαράμ. Δυστυχώς βλέπουμε ότι υπάρχει βία φορές και χωρίς λόγο. Η Νιγηρία πρόσφατα ανακηρύχθηκε μεγαλύτερη οικονομία στην Αφρική. Ακούμε να υπάρχουν ανισότητες στην Ιγυρία ανάμεσα στο βορρά και το νότο, ε, μεγάλη έλλειψη εμπιστοσύνη απέναντι στην κυβέρνηση ε, και γι' αυτό το λόγο οι άνθρωποι δεν αισθάνονται ότι προστατεύονται. Ε, μια μεγάλη διαμαρτυρία της κοινωνίας των πολιτών αφορά την έλλειψη κυβερνητικής αντίδρασης. Έτσι λοιπόν εμείς στηρίζουμε τις ενέργειες που ανέλαβε μια σειρά κυβερνήσεων για να βοηθηθεί η περιοχή Τσιμπόκ, αλλά θέλουμε να υπάρχει πιο συντονισμένη πράξη από την κυβέρνηση της σε συνεργασία με κυβερνήσεις άλλων κρατών. Επόμενος ομιλητής, Μακάβαν, η κυρία Μακάβαν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχουν περάσει 100 περίπου ημέρες από τότε που εξαφανίστηκαν τα κορίτσια και νομίζω σήμερα θα πρέπει να υποσχεθούμε ότι θα συνεχίσουμε την εκστρατεία μας για τα κορίτσια μέχρι να αφαιθούν ελεύθερα και θα αφήσουμε το θέμα να φύγει από τους επιχαίους τίτλους. Συμφωνώ με την κυρία Λάμπερτ ότι πρέπει να συνεργαστούμε με την κυβέρνηση της αλλά και μεταξύ μας να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ε, και ακόμα περισσότερα ε, στους στόχους της χιλιετίας είπαμε ότι κάθε παιδί πρέπει να έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση. Στην Ιγυρία όμως έχουν κλείσει πολλά σχολεία λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων. Η διεθνή κοινότητα πρέπει να τηρήσει τους στόχους της χιλιοτίας. Τα ασφαλή σχολεία είναι ένα κομμάτι όλων αυτών που συζητάμε. Και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να φερθώ στη δουλειά του Gordon Brown και τη γυναίκα του να τους επενέσω. Έχουν αναλάβει πάρα πολλές πρωτοβουλίε για τα ασφαλή σχολεία. Και αυτά πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα ε, της ε, ε, μερίσιας διάταξής μας. Η UNICEF μας ανέφερε ότι στο τέλος του έτους ε, θα έχουμε 25 χρόνια από τότε που γράφηκε η Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Παιδιών. Εμείς εδώ πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε όλα τα παιδιά να έχουν το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Ε, πρόεδρος. Παρακαλώ. Προσπαθήστε συναδελφοί να καθίσετε με ησυχία. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Σένρα Ροντρίγκε για ένα λεπτό. Κυρία Σένρα, έχετε ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ για άλλη μία φορά. Η μία ιδεολογία ή στο όνομα κάποιες θρησκείας ε, δείχνει κάποιος την, ε, το πραγματικό του πρόσωπο και αυτή τη φορά με άσκηση βίας κατά γυναικών, κατά κάποιων κοριτσιών το μόνο τους έγκλημα ήταν ότι ήθελαν να πάνε στο σχολείο όπως έχουν δικαίωμα. Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωσή τους. Απαιτούμε να δοθούν εξηγήσει ότι αυτά τα κοριτσάκια μπορούν να πάνε στο σχολείο. Και αυτά τα κοριτσάκια και όλα τα κοριτσάκια. Θεωρούμε ότι για άλλη μία φορά πάντα σε συγκρούσεις, σε πολέμους, είναι ε, βραβείο, είναι σαν ε, νόμισμα ανταλλακτικό, οι γυναίκες. Οπότε θα πρέπει τα θεσμικά όργανα και η κοινωνία να προσπαθήσουν περισσότερο όσον αφορά τον αγώνα για ισότητα. Να εγγυηθούν τα δικαιώματα των γυναικών σε όλο τον κόσμο και σε όλες τις περιστάσεις. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχουν οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων. Κυρία Γκαμπριέλ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αυτό. Μην αγουστρούμε το σημερινέ αφέ, η βία και οι επιθέσει πρέπει να σταματήσουν. Αυτέ οι ανήλικε και οι ανήλικοι που έχουν απαχθεί πρέπει να απελευθερωθούν. Πρόκειται αυτό για μια τρομοκρατική ομάδα, πρόκειται για την Boko Χαράμ, αλλά το θέμα είναι να πάρουν το μήνυμα και οι Νιγηρινέ αρχέ, γιατί ε, αυτό είναι ένα σύμπτωμα τη δυσλειτουργία του Νιγηρινού κράτου. Υπάρχει ευρύτερο πρόβλημα και θα πρέπει να κάνουμε δύο άξονε για τι δράσει μα. Πρώτα-πρώτα να υπάρχει μεταρρύθμιση όσον αφορά την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη. Και έτσι θα πρέπει οι νιγηριανέ αρχές να μπορέσουν να καταπονεμήσουν την τρομοκρατία σε να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο. Δεύτερο άξονα η περιφερειακή συνεργασία. Γιατί γνωρίζουμε ότι μέρος της χρηματοδότησης τη οργάνωσης αυτής προέρχεται από εμπόριο όπλων, ναρκωτικών και δουλεμπόριο και ότι έχουν τα, τα τους στις ε, γειτονικές χώρες. Επομένω, θα πρέπει ε, σήμερα η, η Αφρικανική Ένωση να λάβουν δράση, να υπάρχει διεθνή συνεργασία. Είναι πιο σημαντικό από ό,τι στο παρελθόν γιατί υπάρχει ε, απειλή από την Μποκ Χαράμ σε όλη την περιοχή. Φέρτε πίσω τα κορίτσια. Γκόμες. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει εδώ σχέση μεταξύ της Μποκοχάραμ και άλλων τρομοκρατικών συμμοριών. Άρα εδώ σοβεί μια ανθρωπιστική κρίση. Έχουμε 2.000 άμαχους που έχουν φωνευθεί σε περίπου 90, 50 επιθέσεις. Άρα υπάρχει εδώ πέρα η ανθρωπιστική κρίση και θα πρέπει επομένως ε, να εμπλακεί εδώ και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Θα πρέπει να γίνει εδώ μια έρευνα με τη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Νιγηρία να κάνει ό,τι μπορεί για να προστατεύσει τον λαό από αυτές τις επιθέσεις. Πρόκειται για κάποιες ε, ανήλικες οι οποίες έγιναν στόχος της Μπόκο Χαράμ. Υπάρχει βέβαια γενικευμένη διαφθορά και στις δυνάμεις ασφαλείας και στις ενόπλες δυνάμεις. Καταπατούνται τα θεμελιώδη δικαιώματα του πληθυσμού, σοβεί φτώχεια, αλλά υπάρχει και βία στη χώρα. Θα πρέπει επομένω η ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ιγυρία να συσχετιστεί με την ε, αντιμετώπιση των προσλημάτων που είναι η αιτία της δράσης της Μπόκο Ο κύριος Μπέλτερ για ένα λεπτό. Κύρια Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Οι ρίζες του κακού στην ε, Νιγηρία είναι πολύ βαθιές. Αυτό το μήνα έχει λαιλατήσει και δολοφονήσει πολλούς αθώους η με έχει κάψει χωριά, έχει στραφεί κατά μάχων Μερικά από αυτά τα μαθαίνουμε, αλλά υπάρχουν και οι, λεγόμενοι σιωπηροί φόνοι, εις βάρος χριστιανών ή πιστών διαφορετικών ε, προσανατολισμών ή δογμάτων, που δεν βρίσκουν θέση στα εφημερίδες και στις ειδήσει έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική οργάνωση η Μπόκο Χαράμ. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνω έκκληση στο Συμβούλιο κατεπηγόντως και με ιδιαίτερη έμφαση να απευθύνει έκκληση στις αρχές της Νιγηρίας και να τους υπενθυμίσει και την ευθύνη τους απέναντι στην κοινότητα των χριστιανών της Νιγηρίας. Διότι δεν υπάρχει καμία δημόσια ενίσχυση, δεν υπάρχει καμία προστασία επαρκής για τους χριστιανούς ε, έναντι των επιθέσεων της Ποκοχαράμ. Απευθύνω λοιπόν έκκληση στους, στις αρχές της Νιγηρίας να μην εγκαταλείψει τους χριστιανούς στη μοίρα τους και να τους προσφέρει κατάλληλη προστασία. Ε, ευχαριστώ κύριε Μπέλτερ. Δέχεστε μία μπλε κάρτα με τη διαδικασία αυτή από τον κύριο Σαρνέτσκι. Κύριε Πρόεδρε, έχω μια ερώτηση προς τον κύριο Μπέλτερ. Και είναι η Θεωρεί ότι ενδεχόμενες κυρώσεις εις βάρος της κυβέρνησης της Νιγηρίας θα μπορούσαν να την ενισχύσουν τελικά στον αγώνα της κατά τον ε, του κίνηματος της Μποκοχαράμ, του Τρομοκράτου της Μποκοχαράμ, γιατί εγώ έχω την πεποίθηση ότι δεν θέλει να τους, ε, να τους καταπολεμήσει. Ευχαριστώ πολύ. 30 δευτερόλεπτα κύριε Μπέλντερ. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Σαρνιέσκη. Έχετε δίκιο απολύτως. Πρέπει να εκφράζουμε βαθύτατη ανησυχία σε σχέση με τη στάση των αρχών της Νιγηρίας, διότι βλέπουμε από έγκυρες πηγές ότι οι αρχές διατήρησης της τάξης, ο στρατός εν ολίγης, έχει ε, διαβρωθεί από στελέχη της Μποκοχαράμ. Και πλέον οι χριστιανοί της Νιγηρίας δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στις ε, δυνάμεις διατήρησης της τάξης, γενικά στις αρχές της Νιγηρίας. Απευθύνω λοιπόν έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ανάληψη ε, αποφασιστικών κυρώσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ τους συναδέλφους όσο το δυνατόν πιο ήσυχα για να συνεχιστεί η συζήτηση. Κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίκα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και εγώ συμφωνώ με την καταδίκη για την απαγωγή αυτών των κοριτσιών από το σχολείο στο Τσίμπο μια φορά σεξουαλική βία. Χρησιμοποιείται αυτό ως ε, όπλο πολέμου. Και πρόκειται για φονταμενταλιστές, πρόκειται για ε, αυτού του είδους πάλι που γίνεται στην Ιγυρία. Αλλά πέραν αυτών, εγώ θέλω να προβληματιστώ και με κάτι άλλο. Το 2013 ήταν η Ιγυρία η πιο πλούσια χώρα, πιο μεγάλο έπειχε από την Νότιο Αφρική. Έχουν πετρέλαιο, έχουν τηλεπικοινωνίες, έχουν βιομηχανία, αλλά το 60% ζει με ένα δολάριο την ημέρα. Αυτό φέρνει απελπισία και αυτό τροφοδοτεί τους εξτρεμισμούς. Άρα βεβαίως θα πρέπει να καταδικάσουμε την Ποκοχαράμ αλλά επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι μια τόσο πλούσια πόλη θα πρέπει να δούμε γιατί βρίσκεται στη θέση 153 του καταλόγου του σχετικού του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει επομένως να δοθούν και κάποιες λύσεις γιατί όλα αυτά τα προβλήματα η απελπισία κάνει τον κόσμο να μην έχει τίποτα να χάσει και να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Φυσικά απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση αυτών των κοριτσιών. Η κυρία Χάουτα το λόγο για ένα μισή λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, οι μαθήτριες του σχολείου της ΣΥΜΠΟΚ είναι ένα σύμβολο του, της φρικαλαιότητας για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται γυναίκες και κορίτσια σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν ε, ό,τι μπορούμε για να προστατέψουμε τα κορίτσια αυτά. Όπως η Μαλάλα στο Πακιστάν η οποία έπεσε θύμα των ε, Ταλιμπάν ε, δολοφονικής επίθεσης. Επέζησε όμως και αυτές τις μέρες βρίσκεται στην Ιγυρία για να ζητήσει από τον πρόεδρο Good luck Jonathan να κάνει ό,τι μπορεί για να φέρει πίσω τα κορίτσια αυτά τα, οι μαθήτριες αυτές ε, του Σιμπόκ έχουν ε, κάθε δικαίωμα στην προστασία μας και πρέπει και εμείς να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να τις φέρουμε πίσω συνθήκες ασφάλειας. Ιδιαίτερα ενισχυτικό όμως ως προς τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών είναι το πρόβλημα της γενετήσης ελευθερίας που καταστέλλεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας μαζί με τη διεθνή κοινότητα ώστε να εξασφαλιστεί το δικαίωμα της επιλογής για το ίδιο της το σώμα από την κάθε γυναίκα, από το κάθε κορίτσι. Να μην αντιμετωπίζονται ως ε, αντικείμενα και ως ε, σκλάβες του σεξ ε, χωρίς καμία αξιοπρέπεια. Πρέπει να παραμείνουν τα φώτα του ενδιαφέροντος διεθνής κοινότητας πάνω στην Ιγυρία μέχρι να αποφυλακιστούν, μέχρι να απελευθερωθούν αυτές οι μαθήτριες. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ να κάθεστε ήσυχα για να μας επιτρέψετε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Οι συνάδελφοι στα πίσω να παρακαλώ να καθίσουν. Και τώρα, κοράω Ιγνάτσιο. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Κοιτάξτε, στις αρχές του 2014 η τζιχαντιστική ε, τρομοκρατική οργάνωση Μποκοχαράμ ε, ε, διέπραξε πάρα πολλούς φόνους ε, ε, και αυτό οφείλεται κυρίως στην παραγωγή του πετρελαίου. Οι περισσότεροι πολίτες στην Ιγυρία ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Σε τίποτα δεν βοήθησε η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ειρήνη και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η τρομοκρατική οργάνωση ενισχύθηκε και η οικονομική κατάσταση της χώρας επιδεινώθηκε. Πάρα πολλές φορέ. βλέπουμε στοιχεία ότι το 2009 γεννήθηκε Μπόκο Χαράμ, αλλά προέκυψαν και οι παρεμβάσεις στη Λιβύη και σε άλλες χώρες. Ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ένοπλες σειράξεις στην Αφρική. Ε, Υπάρχουν οργανώσεις ε, όπως ε, το, ε, οργανώσεις που βοηθούνται από αλλοδαπά trust fund. οφείλουμε να παρέμβουμε για να παρεμποδίσουμε αυτή την αιματοχυσία. Να προσπαθήσουμε να σπάσουμε ε, τις διασυνδέσεις αυτής της ε, τρομοκρατικής οργάνωσης της Boko Haram. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Συναδεινός παρακαλώ και η Ελλάδα μια ευρωπαϊκή χώρα διαφέρουν σε πολλούς τομείς. Ομοιάζουν όμως ως χώρες το εύρος της διαφθοράς, των πολιτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Οι κεντρικές τους κυβερνήσεις είναι ανάλγητες προς το λαό και παρανομίες βουλευτών και υπουργών με τη συνεργασία των πολιτικών κομμάτων δεν οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Στην Ιγυρία η δράση των οργανώσεων Μπόκο Χαράμ και Ανσαρού αποσανατολίζει την κοινή γνώμη από τα πραγματικά προβλήματα. Οι τρομοκρατικέ επιθέσει ρίχνουν στάχτη στα μάτια του λαού το δίθεν πρότυπο ανάπτυξη και τα στα πραγματικά προβλήματα με σκοπό την επιβίωση των πολιτικών και την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων. αναρωτιέμαι όμω είναι δυνατόν το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο να διαφορεί για παρανομίε εντό των κρατών μελών του και να ασχολείται με τη γειτονιά του. στην ελλάδα η συγκυβέρνηση εξυπηρετώντα ιδιωτελεί σκοπού με τη συνδρομή τη εκτελεστική και δικαστική εξουσία έχει εγκαθιδρύσει μια ιδιότυπη δικτατορία. στην ελλάδα δεν υπάρχει μπόκο χαράμ και ανσαρού υπάρχουν επίουρκοι δικαστικοί διεφθαρμένη πολιτική χρηματισμός κρατικών παραγόντων και πολιτική δίωξη αντιπάλων. έτσι ο γενικός γραμματέας και οκτώ βουλευτές της χρυσής αυγής της τρίτης πολιτικής δύναμης οδηγήθηκαν στη φυλακή με προσχηματικές κατηγορίες κατά εντολή του πρωθυπουργού σαμαρά. σε αριθμό βουλευτών κατά παράβαση του άρθρου 19 του οηε αντισυνταγματικά έχει απαγορευτεί η ελευθερία γνώμης και Ευχαριστώ

Κύριε Πρόεδρε, έχουμε αυτό το ψήφισμα του Κοινοβουλίου όσον αφορά την κατάσταση αυτή στην Ιγυρία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το υποστηρίξουμε γιατί πρόκειται για αυτή την τρομοκρατική οργανώση την Μποκό Χαράμ, η οποία όχι μόνο έχει ε, ε, σκοτώσει κόσμο, αλλά έχει χτυπήσει και τον πολιτισμό και την παιδεία. Έχουμε όλα αυτά τα κοριτσιά τα οποία ε, απήκθησαν και που σκλάβε. Αυτό αυτό έχει κάνει το γύρο του κόσμου και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προσέξτε, δεν είμαστε μόνο ευρωβουλευτέ, αλλά είμαστε και γονεί και ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι τα παιδιά. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, τόσο ώστε τα παιδιά αυτά να γυρίζουν σπίτι του. Και οπότε θα χρειαστεί αποφασιστική δράση, αλλά και συνεργασία με την Νιγηριανή κυβέρνηση, με τον ΟΗΕ, με την ε, Αφρικανική Ένωση. Επίση, θα πρέπει να βοηθήσουμε και τι οικογένειε των ε, απαχθισών. Τώρα, όσον αφορά τα μακροπρόθεσμα μετά που θα πρέπει να λάβουμε, θα πρέπει με συστηματικό τρόπο να βοηθήσουμε τόσο σώστη χώρα να αποκτήσει σταθερότητα. Σας ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρος, κυρία Κέντζε. Κέντζε. Signora Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, στη συζήτηση βλέπουμε ότι υπάρχει μημάτια όσον αφορά την φτώχεια. Αυτή είναι η ρίζα της φτώχειας. Ε, αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν είναι τυχαίο κυρία Πρόεδρε ότι η Μπόκο Χαράμ ε, μεταφράζεται με τους εξής τρόπους ότι είναι κρίμα να υπάρχει δυτική εκπαίδευση όπως ε, και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι γυναίκες δεν έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση, το οποίο είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Δεν είναι βέβαια αυτός σκοπός, αλλά αυτός είναι ο δρόμος για να μπορεί κανείς να ασκήσει και τα άλλα του δικαιώματα. Και ε, πρέπει να ταχθούμε υπέρ όλων των πράξεων που θα οδηγήσουν στο να επιστρέψουν στα σπίτια τους τα κορίτσια. Να πάψουν να υπάρχουν αυτές οι τρομοκρατικές ενέργειες της Μπόκο Χαράμ. Κύριε Πρόεδρε, εγώ προτείνω για το 2014 υποψηφιότητα ε, για το βραβείο Σαχάροφ να είναι οι μητέρες αυτών των κοριτσιών που απήχθησαν να επαναφέρουμε, να φέρουμε πίσω τα κορίτσια μας. Bring back our girls. Αυτό θα πρέπει να είναι το σύνθημά μας. Κυρία Ντότς, έχετε ένα λεπτό στη διάθεσή ναι. σας. One. Mm. Το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Με χαρά συμμετέχω στη συζήτηση σήμερα και βλέπω ότι επικεντρωνόμαστε σε εκείνους οι οποίοι ε, ταλαιπωρούνται από τις διώξεις λόγω θρησκείας. Η περίπτωση όμως των κοριτσιών της ε, Νιγηρίας είναι κάτι περισσότερο από ανησυχητική. Έχουμε ρίξει τα φώτα του ενδιαφέροντος διεθνούς κοινότητα στην κατάσταση των ε, ε, κατοίκων στη νότια Νιγηρία, χιλιάδων χριστιανών που υποφέρουν από τις επιθέσεις της Μποκοχαράμ. Στο τελευταίο κοινοβούλιο, μαζί με τον συνέλφο Μπέλντερ, υποστήριξα του Χριστιανού και τι βόρείε. Νιγηρία προσκαλέσαμε μάλλον χριστιανού τη βόρεια Νιγηρία στο κοινοβούλιο. Ένα από αυτού ε, μας αφηγήθηκε πω ήρθε μια ομάδα της Μποκοχαράμ στο σπίτι του, του έβαλε ένα μαχαίρι, ένα όπλο στο κεφάλι και του είπαν ε, ότι πρέπει να αλλάξει θρησκεία. Αρνήθηκε όμως ο συγχωριανός αυτός και ε, τον πυροβόλησαν στο πρόσωπο. Επεβίωσε όμως. Ζήτησε από τη γυναίκα του να τρέξει, να φωνάξει τους γείτονες ότι έρχεται η Μπόκο Χαράμ και να κρυφτούνε. Όταν γύρισε πίσω η γυναίκα του, του ε, τον ενημέρωσε δεν είχε μείνει κανεί ζωντανό στο χωριό. Ήταν ο μόνο ο οποίο είχε μείνει ζωντανό από θαύμα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε το θάρρο στο Κοινοβούλιο να καταγγέλουμε τι ε, διώξει όλων αυτών των αθών για λόγου μόνο θρησκεία. Σα ευχαριστώ πολύ. Ο κατάλογος των ομιλητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων έχει ολοκληρωθεί. Έχουμε τώρα τη διαδικασία Catch the Eye και παρακαλώ να αντισεβαστείτε αυστηρά την, ε, τη διάρκεια του ενός λεπτού που δίνουμε. Ο κύριος Ταραμπέλα, πρόεδρε τις τελευταίες εβδομάδες, έχει αναπτύξει διάφορες δολοφονικές επιθέσεις σε χωριά της Νιγηρίας, η Η τρομοκρατική οργάνωση Μπόκο Χαράμ, επιθέσεις οι οποίες συμπληρώνουν την ε, φαιά εικόνα, ζωφερή εικόνα της ε, απαγωγής πάνω από 200 κοριτσιών στην περιοχή Σιμπόκ Μπορνό της Νιγηρίας. Η κατάσταση παρά τις πολλές προσπάθειες κατάσταση παραμένει πολύ αβέβαιη και φοβόμαστε για το χειρότερο καθημερινά. Καταδικάσουμε λοιπόν βεβαίω όλε αυτέ τι ακρότητε, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να επιβεβαιώσουμε την υποστήριξή μα στην κυβέρνηση τη Νιγηρία, ώστε να μπορέσει εκείνη πραγματικά να αγωνιστεί κατά τη Μποκοχαράμ, κυρίω με την αποστολή διπλωματών από πλευρά μα, αλλά και με μια στρατιωτική, εστιασμένη στρατιωτική ε, υποστήριξη για να καταπολεμηθούν αυτοί οι αντάρτε, τρομοκράτε. Πρέπει να ενώσουμε πάνω από όλα όμω τη φωνή μα ότι ποτέ δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό το απαράδεκτο. Ένα λεπτό παρακαλώ. Mr. Κύριε Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Μποκο Χαράμ, ε, μεταφρασμένη λέξη, σημαίνει ότι τα βιβλία και η παιδεία είναι αμαρτία. Προηγουμένως ε, είπε κάποια συνάδελφος ότι ε, ο πατριαρχισμός ε, δείχνει το πρόσωπό του. Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό. Το ακραίο Ισλάμ δείχνει το πρόσωπό του. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με μία από τις πλέον ακραίες Ισλαμιστικές οργανώσεις που υπάρχουν στον κόσμο και στην Ιγυρία. Υπάρχουν όμως και σε άλλες χώρες αυτές οι οργανώσεις. Τα εγκλήματα αυτών των ομάδων τους τελευταίους μήνες εμφανίστηκαν σε επιχαίους τίτλους στις εφημερίδες. Πολλοί συνάδελφοι τα ανέφεραν αυτά και αυτή η οι τίτλοι προκαλούν φόβο. Ε, είναι ε, γεγονότα που μας κάνουν να τριχιάζουμε. Έχουμε 300 κορίτσια που απήχθησαν. Στις αρχές του Ηλίου σφαγιάστηκαν 60 άνθρωποι. Αυτές είναι οικογενειακές ε, τραγωδίες και δεν νομίζω ότι μπορούμε να τις προβάλλουμε εδώ με το σωστό τρόπο. Αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι πραγματικά η χειρότερη μορφή του Ισλάμ και θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να το καταδικάσουμε με τον πιο αποφασιστικό τρόπο επόμενη μιλήτρια, η κυρία Οντεμπερκ. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ αυτές οι βίες επιθέσεις της ε, Μπόκο Χαράμ στη Βόρειο Νιγηρία οδηγούν σε αποσταθεροποίηση ολόκληρης περιοχής. Από το 2010 διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν επιθέσεις κατά των θεσμών, κατά των σχολείων, ε, δολοφονούνται άνθρωποι, πολλά παιδιά, κατόπιν ακολούθηση απαγωγή 200 ε, κοριτσιών από το σχολείο τους που βρίσκονται σε άγνωστο μέρος. Το Μπόκο έχει οδηγήσει σε ανθρωπιστική κρίση και αυτή έχει επεκταθεί και στις γειτονικέ χώρες. Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις, να αντιμετωπιστεί η ανεργία. Για να γίνουν όλα αυτά χρειαζόμαστε ισχυρούς θεσμούς. Πρέπει να εμφυσίσουμε ασφάλεια στους πολίτες έτσι ώστε να μην καταστούν θύματα του ακραίου Ισλάμ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η διαδικασία Catch the Eye ολοκληρώθηκε. Γι' αυτό, συνάδελφοι, ε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να είστε ήσυχοι και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Επίτροπο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρέπει να σας πω ότι συνεχίζουμε να ανησυχούμε για την κατάσταση στην Ιγυρία. Στην Ιγυρία όπου συνεχίζονται οι βίαιες επιθέσεις που συνεχίζουν να τρομοκρατούν τους πολίτες. Η ύπατη εκπρόσωπος, η κυρία Άστον, καταδίκασε απερίφραστα την ε, δολοφονία χωρίς κανένα κριτήριο εκατοντάδων πολιτών και την απαγωγή πάνω από 200 κοριτσιών στο Μπόρνο. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε να ζητάμε την ε, απελευθέρωση των κοριτσιών αυτών χωρίς καμία προϋπόθεση. Επίσης ζητάμε οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν στα δικαστήρια. Οι σκέψεις μας είναι στις οικογένειες των κοριτσιών που επιθυμούν διακαώς τα κορίτσια τους να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Ξέρετε, αν δεν κάνετε ησυχία, ούτε καν εγώ δεν ακούω τη φωνή μου, λέει η Επίτροπος. Η βία στην ε, Νιγηρία διακόπτει η πρόεδρος με συγχωρείτε κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να σας ε, παρακαλέσω θερμά ε, να ε, κάνουμε ησυχία για να δώσουμε δυνατότητα στην κυρία Επίτροπο να μιλήσει και να συνεχίσουμε τη συζήτηση γιατί εντός ολίγου της χαλιώς πρέπει να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Η Επίτροπος. Η βία λοιπόν στη Νιγηρία έχει επιδεινώσει τη ζωή των πολιτών από το 2009 Μιλάμε για περίπου 5.000 χαμένες ζωές, ε, μιλάμε για περίπου 500.000 εκτοπισμένους, για την καταστροφή εκατοντάδων σχολείων και κυβερνητικών κτηρίων. Ε, μία αδύναμη οικονομία βόρειο-ανατολικά επιδεινώθηκε περαιτέρω και αυτό που ανισχύει περισσότερο είναι ότι από τις αρχές του έτους οι επιθέσεις αυτές λαμβάνουν χώρα σχεδόν κάθε μέρα και από τον Ιανουάριο μόνο ε, μιλάμε για 1.500 μέχρι 2.000 αθώους ανθρώπους οι οποίοι δολοφονήθηκαν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέταξε την Μπόκο Χαράμ τον περασμένο μόλις μήνα ως τρομοκρατική οργάνωση μία μόλις ημέρα μετά την καταδίκη αυτής της οργάνωσης ε, από τα Ηνωμένα Έθνη. Απαράδεκτες λοιπόν εγκληματικές ενέργειες αυτής της οργάνωσης κατά τόσο χριστιανών όσο και μουσουλμάνων. Τα αίτια της ε, βίας ε, και η ίδια η βία θα συνεχιστούν και θα συνεχίσουν να στιγματίζονται από το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο, το οποίο νέο ναι, αυτό ταμείο θα εστιάσει την προσοχή του κυρίως στο βορρά της χώρας, προσφέροντας υποστήριξη στον τομέα της και της ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρούσα στην Ιγυρία και με ανθρωπιστική βοήθεια προσφέροντας 5 εκατομμύρια ευρώ στα βόρεια-ανατολικά κράτη, κυρίως εν είδη αντίδρασης ε, της ε, κρίσης ε, τροφίμων. Σε πολιτικό τώρα επίπεδο, τα ανθρώπινα δικαιώματα παραμένουν απόλυτη προτεραιότητα των σχέσεών μας με την Ιγυρία και περιλαμβάνονται στους τακτικούς υπουργικούς διαλόγους. Οι καταχρήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από το στρατό της Νιγηρίας πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω και όσοι φέρουν ευθύνη να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την κυβέρνηση και το λαό της Νιγηρίας στον αγώνα της κατά της τρομοκρατίας και της βίας για την υπερίσχυση του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συνεργαζόμαστε με τις αρχές της Νιγηρίας για να υπάρξει ένα τέλος σε αυτό τον κύκλο της βίας μέσα από πολλές ενέργειες συμπεριλαμβανομένου και του συνεχούς πολιτικού διαλόγου ε, με στοχευμένες πράξεις ε, που θα έχουν ως αντικείμενο την καταπολέμηση των αιτίων της ρίζας της βίας. Ε, πρόεδρος. Τώρα. επιλήξει συζήτηση.